Uh, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρο. αρχίζουμε με το σημείο 14 της ημέρησης που Θα συμπροεδρεύσουμε τον κύριο Γκουαλτιέρη, τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και το θέμα μας είναι ο έλεγχος των διαθεσίμων ρευστών που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προεισαγωγικά Καλώ όρισαν οι συνάδελφοι της Οικονομικής Επιτροπής και πάλι για άλλη μια φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που δύναμη του άρθρου 55 του κανονισμού συνεργαζόμαστε για κάποιο νομοθέτημα και η κάθε επιτροπή συμβάλλει. Πολύ σημαντικό το θέμα είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και αυτά τα συζητήσαμε και τα ακούσαμε από τον Επίτροπο με το χαρτοφυλάκιο τη ασφάλεια. Οπότε θα παίρνουμε κάποια μετώπιση να σταματήσουν αυτέ τις δραστηριότητε και να σταματήσει η εκμετάλλευση από πλευρά των ε, εγκληματιών τη καταστάσεως. Αυτό είναι ο στόχος μας και τώρα να δώσω τον λόγο στον Ρομπέρτο Γκολτιέρη, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του πρόκειται να να παρουσιάσει την συνάντησή μας. Ευχαριστώ Κλόντεφ και είναι για μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε εδώ και έτσι ξεκινούμε ακόμα μια προσπάθεια δυνάμη του άρθρου 55 σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Δημοκρατικών Ελευθεριών διότι ήταν πολύ αγαστή συνεργασία μας για το ξέλιμα του χρήματο και πιστεύουμε ότι και άλλη μια φορά θα είναι παραγωγική συνεργασία μας για αυτό το τόσο σημαντικό νομοθέτημα που αφορά τη, τη, τον έλεγχο αυτών των ροών μετρητών ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι θα καταπολεμήσουμε το, το, την, την φοροδιαφυγή, την τρομοκρατία, το ξέρουμε χρήματος, οπότε αμελητή ας αρχίσουμε και έχουμε αυτό το αξιόλογο σχέδιο κειμένου. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ρομπέρτο και τώρα να δώσουμε το λόγο στον συνεισηγητή της Επιτροπής Λίμπες, τον κύριο Λόπες Αγγιλάρ. Φερνάντο, έχεις πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε Μωράστη, κύριε ε, τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας ε, παρουσιάσω το σχέδιο της έκθεσης σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των ευθών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ τράτω με τις ευκαιρίες για να ευχαριστήσω και την ε, γραμματεία που διοργάνωσε αυτή την κοινή συνεδρίαση, δηλαδή από κοινού με μέλη των δύο επιτροπών έκονα και ΛΥΜΠΕ που συνεργάζονται σε σχέση με αυτόν τον φάκελο προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της καταπολέμησης τρομοκρατία ε, και ειδικότερα τη χρηματοδότηση αυτή εγκληματικών δηλαδή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την τρομοκρατία, αλλά και άλλε μορφέ σοβαρού διασυνοριακού εγκλήματο. Ε, βρισκόμαστε δηλαδή στην απαρχή μια ε, πολύ καλή συνεργασία που έχει ξεκινήσει μεταξύ των δύο επιτροπών, ΛΥΜΠΕ και ΕΚΟΝ. Πολύ καλή συνεργασία και με την κυρία Ντελβό, την συνεισηγήτρια, η οποία θα πάρει το λόγο και μετά από μένα. Στο πλαίσιο βέβαια ε, των αρμοδιοτήτων της ε, κάθε κοινοβουλευτική Επιτροπής και της ε, κάστοτε από τις δύο ομάδες, ούτως ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην εκπόνηση της έκθεσης και να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Η καταπολέμηση λοιπόν της τρομοκρατίας και του εγκλήματος είναι το γενικότερο μας πλαίσιο και κατά συνέπεια τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ώστε να σταματήσει η χρηματοδότησή τους. Έχουμε δηλαδή διαφορετικούς ε, κανόνες που ισχύουν σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, των ρευστών διαθεσίμων και οι οποίοι θα αναθεωρηθούν τώρα στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, μέσω δηλαδή κατάργησης ενός εφιστάμενου κανονισμού. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μία ε, πανευρωπαϊκή προσέγγιση σε ό,τι αφορά τον έλεγχο ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται αλλά και εξέρχονται στην Ένωση προκειμένου να εγγυηθούμε την εύρυθμη λειτουργία τη ε, κοινή αγορά αλλά και προκειμένου να εγγυηθούμε την προστασία των πολιτών μα αλλά και των επιχειρήσεών μα. Ε, και βέβαια εδώ οι τελωνιακέ αρχέ βρίσκονται στην αιχμή του δόρατο γιατί αυτέ που είναι αρμόδιε τόσο για τον έλεγχο των επιβατών αλλά και για την κυκλοφορία εμπορευμάτων και αποστολών. Η ε, συνεργασία λοιπόν μεταξύ αυτών των ελληνικών αρχών θα πρέπει να επιταθεί προκειμένου να αποφύγουμε την ε, ε, παράκαμψη από την πλευρά των εγκληματιών αυτών των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Δεκέμβριο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβησε μια πρωτοβουλία με την υιοθέτηση ενό πακέτου μέτρων προκειμένου να εφαρμοστεί ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο σε ό,τι αφορά το ξέπλυμα βρωμικού χρήματο, τι ροέ χρημάτων αλλά και την δέσμευση και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και Βέβαια, αυτή η πρωτοβουλία ε, λαμβάνει η χώρα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που αναλάβαμε στο πλαίσιο του σχεδίου δράση για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και τη ε, χρηματοδότηση τη τρομοκρατία το Φεβρουάριο του 2016. Έτσι λοιπόν, έχουμε μπροστά μα μία πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την βελτίωση του κανονισμού σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των ρευστών διαθεσίμων που είχε ε, τέθει σε ισχύ το 2005 για τον έλεγχο λοιπόν των ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται και εξέρχονται στην Ένωση. Ε, ποια είναι η νομική βάση του άρθρο 114 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, που στοχεύει στην προσέγγιση, στην αμοιβαία προσέγγιση των εθνικών διατάξεων των κρατών μελών προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργία της νέας αγοράς αλλά και το άρθρο 33 που προβλέπει την ενίσχυση της συνεργασίας των τελωνιακών αρχών των κρατών μελών αλλά και μεταξύ των τελωνιακών αυτών αρχών και της Επιτροπής. Οι προτάσεις που κάνει τώρα για αλλαγή η Επιτροπή ε, είναι να γίνουν αυστηρότεροι οι έλεγχοι ε, των ατόμων που εισέρχονται, εξέρχονται από την Ένωση ε, και έχουν μαζί τους τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Αυτό είναι το κατώτατο λοιπόν όριο. 10.000 ευρώ είτε σε ρευστά είτε σε πολύτιμα αγαθά τα οποία αποστέλλονται και μέσω ταχυδρομικών δεμάτων ή εμπορευματικών αποστολών. Ο στόχος είναι να οι αρχές να μπορούν να αναλαμβάνουν δράση ακόμα και σε περιπτώσεις όπου ε, τα μεταφερόμενα αυτά ρευστά διαθέσιμα βρίσκονται κάτω από το κατώτατο όριο των 10.000 ευρώ, όπου υπάρχει υποψία για κλιματική δράση και προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών και ε, επιτροπής. Ε, επίσης, ειδικότερα δηλαδή, ο ορισμός εδώ των ρευστών περιλαμβάνει πλέον και το χρυσό και άλλα πολύτιμα αγαθά, αλλά και προπληρωμένες κάτες πληρωμές, οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με ένα συγκεκριμένο τραπεζικό ή άλλο χρηματικό λογαριασμό και κατά συνέπεια δεν υπάγονται στην τυποποιημένη μέχρι στιγμή τουλάχιστον ε, τελωνιακή διασάφηση. Άρα λοιπόν αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται πλέον στον ορισμό των ρευστών. Αυτό περιλαμβάνει η νέα πρόταση τη Επιτροπή. Η νέα πρόταση επιτρέπει επίση στι ε, αρμόδιε αρχέ να δεσμεύουν προσωρινά ε, ρευστά διαθέσιμα όταν εντοπίζουν κάποια μεταφορά ρευστών, ακόμα και όταν αυτή είναι χαμηλότερη από την κατώτατη αξία που ανέφερα μόλι τώρα, αλλά υπάρχει υποψία ότι σχετίζεται με κάποια εγκληματική δραστηριότητα. Αυτό δηλαδή δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο του σημερινού κανονισμού. Ο στόχος λοιπόν είναι να ενημερωθεί ο κανονισμό και να ενισχυθεί και το πεδίο εφαρμογή του ισχύοντο κανονισμού. Επίσης η πρόταση της Επιτροπής στοχεύει ε, στην ενιαία, ομοιόμορφη εφαρμογή ε, των ελέγχων μέσω ε, αρμοδιοτήτων ε, με ε, ε, αντίστοιχε εξοδοτήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ισχυθεί η ανταλλαγή των πληροφοριών, να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία. Εδώ δηλαδή το σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών είναι πολύ σημαντικό, αλλά και η μέσω της παροχής πληροφοριών από τα κράτη-μέλη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία ε, τα οποία θα μας εξηγήσει τη συνεισηγήτρια από την ε, Επιτροπή ΕΚΟΝ, την κυρία Ντελβού, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα συνόδευτα μετρητά και πώς αυτά ε, διαφοροποιούνται από τα συνοδευόμενα ρευστά διαθέσιμα, το, ποια είναι η διαφορά για παράδειγμα της αξιολόγησης κινδύνου και τη εκτίμηση κινδύνου και ποιε είναι οι διαδικασίε για την ενίσχυση τη ανταλλαγή πληροφοριών, ειδικότερα μέσω των συστημάτων μηχανοργάνωση, δηλαδή πληροφορική και βέβαια και ο μηχανισμός ε, ε, της ε, Ευρωπαϊκής Μονάδας Οικονομικών Πληροφοριών. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία που πρότεινε η Επιτροπή. Εμείς είμαστε υπέρ του να δοθεί συνέχεια σε αυτή την πρόταση, αλλά από εκεί και μετά προφανώς είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις σε σχέση με αυτή την πρόταση και η κυρία Ντελβό θα συνεχίσει τώρα την παρουσίαση αυτή. Ευχαριστώ ο Πρόεδρος. Κυρία Ντελβό, έχει τώρα το λόγο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έγινε πραγματική συνεργασία και είναι εξαιρετική δουλειά των συνεισηγητών. Ε, οπότε να σας παρουσιάσω αυτό το κείμενο γιατί πρώτα-πρώτα ως διευκρινήσεις προσθέτουμε στο άρθρο 2 έναν ορισμό του έχοντος τα ρευστά, του μεταφέροντος τα ρευστά τέλος πάντων και στο άρθρο 3 συμπληρώνουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την δήλωση ούτω ώστε να μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρμόδιες αρχές. Ε, επίσης, στο άρθρο 8 προτείνουμε μια μείωση της προθεσμίας με στις οποίες οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαβιβάσουν τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ε, δήλωση στην ε, μονάδα οικονομικών πληροφοριών γιατί αν υπάρχει κάποια υποψία θα πρέπει να υπάρχει περιθώριο επιτάχυνση τη διαδικασία. Κατόπιν έχουμε το άρθρο 13 για τι κυρώσει σε περίπτωση αποφυγή, παράληψη τη δήλωση όσον αφορά το ρευστό. Αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα. Αλλά θεωρούμε ότι υπάρχουν σημαντικέ διαφορέ στι εθνικέ ρυθμίσει για τι κυρώσει. Οπότε είπαμε ότι για να σταματήσει ο τουρισμός της επιλογής κράτους μέλους θα πρέπει όλα αυτά να κινούνται στο επίπεδο του 20 έως 40% ως κύρωση επί του συνολικού ποσού που μεταφέρεται. Και επαναλαμβάνω είναι η κύρωση για την αποφυγή δήλωση τόσο ώστε να τιμωρηθούν αυτοί που διαπράττουν το σχετικό αδίκημα. Στο 15 για να μην μπορεί κανεί να διαλέξει από ποια χώρα θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανάλογα με το ποια τον συμφέρει, θα πρέπει οι σχετικέ πληροφορίε που αφορούν ε, τι ε, παραβάσει να είναι κάτι στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί υπάρχει σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών το οποίο λειτουργεί εύρυθμα. Πρώτον το σύστημα τελωνιακών πληροφοριών και θέλουμε να θεσπίσουμε νέα εργαλεία για την ανταλλαγή των πληροφοριών. Δύο λόγια τώρα όσον αφορά τι εκτελεστικέ πράξει και τι κατανάθεση πράξει κατά εξουσιοδότηση και οπότε είπαμε θα πρέπει να γίνει η τροποποίηση του παραρτήματος του σχετικού κανονισμού που ορίζει τι πάει να πει ρευστό, προπληρωμένες κάρτες, επιταγέ κλπ. Διότι θα πρέπει να υπάρχει ταχεία αντίδραση εάν κάτι σκαρφιστούν καινούριο για να διακινήσουν αυτό. Οπότε σύμφωνα με τις κατασκευότητες πράξεις θα πρέπει να δούμε τι έντυπα θα υπάρχουν, τι κανόνες τεχνικοί θα υπάρχουν για την ανταλλαγή πληροφοριών. Όμως τα κριτήρια σε σχέση με διαχείριση του κινδύνου, οπότε υπάρχουν κάποιες υποψίες. Αυτό δεν είναι τεχνικό, τεχνοκρατικό θέμα. Είναι θέμα πολύ σημαντικό και άρα θα πρέπει τα κριτήρια να καθοριστούν με κατανάθεση κατεξοδότηση πράξη και όχι με εκτελεστικές πράξεις. Τέλος, κάτι το οποίο οδήγησε σε προβληματισμό στο Συμβούλιο είναι το τι γίνεται με τα ρευστά τα οποία αποστέλλονται με κάποιο τρόπο είτε με ταχυδρομείο είτε με άλλο τρόπο. Δεν προβλέπεται εδώ δήλωση. Το θέμα είναι όμως ότι θα έπρεπε να θεσπιστεί τέτοια υποχρέωση ακούσαμε τα διάφορα επιχειρήματα, τις επεξηγήσεις. Υπάρχει πρακτικό πρόβλημα για επιβολή τέτοιες δήλωσης. Ποιος είναι υπόχρεος στην υποβολή της, ο αποστολέας ή ο παραλήπτης. Μα μην ξέρει τίποτα. Και ποιανό κράτους οι αρχές θα πρέπει να αναλάβουν τις σχετικές ενέργειες, γιατί ας πούμε μπορεί να μπουν τα χρήματα από άλλη χώρα και όχι σε εκείνη πού είναι ο παραλήπτης. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα προβλέπει ο κανονισμός για την υποχρέωση του. Αλλά υπάρχει έτσι και αυτή η ρήτρα και θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον πρέπει να έχουμε τέτοια υποχρέωση δήλωσης για τα μη συνοδευόμενα ρευστά ε, έχουμε αυτή την προθεσμία της ε, ρέτης ανθεώρησης που ισχύει για τρία χρόνια μετά τη θέση του κανονισμού. Αυτά είναι οι βασικέ αλλαγέ και βέβαια είμαστε πρόθυμοι να τα συζητήσουμε και είμαστε ανοιχτοί, δεν επιμένουμε για κανένα σημείο. Ο πρόεδρος Γκολτιέρη, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να τηρήσετε αυτό το χρονικό των δύο λεπτών για κάθε σκιώδη εισηγητή, ο Φούλιο Μαρτουσέλο, τώρα για την Οικονομική Επιτροπή και για το ΕΛΚ. Ευχαριστούμε. Μπράβο για αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το κείμενο. Και είναι το θέμα αυτών των ρευτών που αφορούν εγκληματικές δραστηριότητες. Και σας υπενθυμίζω ότι έχουμε τώρα κράτος δικαίου, όχι αστυνομικό κράτος. Και άρα θα πρέπει με αυτή την έκθεση να αποφύγουμε να υπάρχουν υπερβολικές, υπερβολικές μονίες στις υποψηφίες και έτσι να μην έχουμε υπερβολή από πλευράς αστυνομίας ή τελωνίων. Και είπαμε ότι το ποσό το οποίο μεταφέρεται πολλές φορές μπορεί να είναι μικρότερο από αυτού που περιχαραγώνει το νομοθέτημα και εδώ είναι το θέμα της υποψίας το κατά πόσον μπορεί αυτό το χρήμα να προέρχεται από κάποιο έγκλημα που διαπράχθηκε και άρα θα πρέπει να υπάρχει κράτος δικαίου και όχι αστυνομικό κράτος. Αυτό είναι ο κίνδυνος. Άρα θα πρέπει να έχουν ακρίβεια οι κανόνες δικαίου και να μην απονέμουν αρμοδιότητες στην αστυνομία, μην απονέμουν ιδιαίτερα μεγάλη διακριτική ευχέρεια και έτσι να διώκεται κάποιος Ευρωπαίος επί τη βάση αυτού του πνεύματος της υποψίας που θέλουμε να κατησχύσει. Έχουμε επομένως αυτό το όριο 10.000, το θέμα είναι αν αυτό θα κατέβει. Έτσι κι αλλιώς να είναι ακριβείς οι ρυθμίσεις. Και ξεκάθαρο το τι κριτήρια θα χρησιμοποιούνται τώρα όσον αφορά την αποθήκευση των πληροφοριών. Πρώτα πρώτα αυτές οι πληροφορίες ε, σώζονται και κρατούνται σε περίπτωση που κριθεί ότι κάποια μεταφορά μετρητών επιδέχεται δίωξη. Τώρα η κάθε χώρα έχει άλλη ρύθμιση και έχουμε πάρα πολλές εμπορικές συναλλαγές και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι ηλεκτρονικής πληρωμής για αυτές. Άρα θα πρέπει να προβληματίσει αυτό και επίσης το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα ηλεκτρονικά νομίσματα όπως τα bitcoin. Γιατί είδαμε ότι και για τη μαφία έχει ε, αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμα αυτά τα νέα νομίσματα και για άλλες εγκληματικές ενέργειες. Και άρα με αυτές τις ε, μεταφορές χρημάτων να μην ε, ωφελείται το έγκλημα. Για το έλστον. Ο κύριος Άντεμος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπροσωπώ τον κύριο Ράντεφ που είναι εισηγητής ε, του ΕΛΚΑ σκιώδης δηλαδή, ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να παρευρεθεί. Τα τελευταία τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, ιδιαίτερα τα μέτρα για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης ε, της ε, τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Οι τροπολογίες ε, επί του κανονισμού για τον έλεγχο των ρευστών διαθεσίμων άνω των 10.000 όταν εισέρχονται και εξέρχονται από την Ένωση επεκτείνεται για να καλύψει εναλλακτικές ε, στο ρευστό χρήμα. Θα βελτιώσει τη συνεργασία λοιπόν για να καταπολεμηθούν και αυτές οι μορφές χρηματοδότησης. Ως και όδης για την πέμπτη οδηγία κατά της ε, νομιμοποίησης προϊόντος εγκλήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σας καλώ να μην υπάρξει σύγχυση μεταξύ των διατάξεων της πέμπτης αυτής οδηγίας με τις διατάξεις του παρόντος κειμένου. Τα κείμενα αυτά είναι συμπληρούμενα. πρέπει λοιπόν να είναι σαφής αυτός ο διαχωρισμός. Ο κύριος Ράντεφ προσβλέπει στη στενή συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών για την περαιτέρω εξέταση του θέματος αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το ECR. Οι στόχοι που προτείνει ο κανισμός αυτός ε, είναι απόλυτα σωστοί. Σε αυτό συμφωνούν ε, φυσικά και όλες οι άλλες ομάδες. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τις ε, απόπειρες των εγκληματιών που προσπαθούν να χρηματοδοτήσουν την εγκληματική του δραστηριότητα μέσω ε, αυτού του χρήματος. Πρέπει να τους σταματάμε στα σύνορα όμως. Τα μέτρα που θα πάρουμε δεν θα πρέπει να θίξουν και τους αθώους που θέλουν να εισέλθουν ή να εξέλθουν στην Ένωση. Τα μέτρα λοιπόν αυτά πρέπει να είναι ανάλογα με τους στόχους τους. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ταξιδεύω συχνά και συχνά πρέπει να συμπληρώσω αυτά τα έντυπα όπου τίθεται το ερώτημα αν πρόκειται να εισέλθω με άνω των 10.000 ευρώ και απαντά όχι. Διερωτώ με πόσοι που έχουν παράνομες προθέσεις και που έχουν πάνω από 10.000 ευρώ στην τσέπη τους λένε ναι. Βάζουν ναι στο κουτάκι. Πώς πιάνουμε με αυτά τα έντυπα. Αν εσείς ε, ξέρετε ότι θα συλληφθείτε θα βάλετε ναι. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν εάν οι στόχοι που επιδιώκουμε επιτυγχάνονται με αυτές τις διαδικασίες και έχω κάποιες αμφιβολίες. Όπως είπε και ο Σάλφος Μαρτουτσέλο, πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε την υποψία να θεωρούνται όλοι ύποπτοι. Πρέπει να ε, περάσουμε από μια διαδικασία που θέτει υπερβολικές ε, απαιτήσει σε όλους προς την αύξηση των αρμοδιοτήτων των τελωνίων που θα πρέπει να βασίζουν την προσπάθειά τους ε, στην ε, ενδεχόμενη ύπαρξη αρχικής υποψίας. Πιστεύω λοιπόν ότι οι προτάσεις που έκανε η Κομισιόν και οι δικές μας είναι θετικές. Χαίρομαι που έχουν διευκρινιστεί κάποιοι ορισμοί και θεωρώ ότι είναι σωστή η προσέγγιση γενικά. Η προσέγγιση δηλαδή ότι δεν θα πρέπει να περιοριζόμεθα σε ρευστό αλλά και σε άλλες μορφές που είναι πολύ κοντά στο ρευστό αλλά εάν ορισμένοι θέλουν, ε, για παράδειγμα, να φοράνε ένα ρόλεξ με διαμαντάκια, δεν θα πρέπει να θεωρούνται κατά ανάγκη υπο... Ή, για παράδειγμα, όταν Θέλουμε κατά κάποιο τρόπο να δούμε ε, ε, εάν σε κάποια αποσκευή έχουν, ε, έχει κρύψει κανείς διαμάντια ή άλλους πολύτιμους λίθους ή αν για παράδειγμα σε κάποια αποσκευή έχουμε κάποιες προπληρωμένες κάρτες αλλά όταν γίνεται ένα ερωτηματολόγιο δεν βέβαια παραδέχεται εκείνος που μεταφέρει αυτές τις κάρτες ότι περιλαμβάνονται στις αποσκευές του. Άρα λοιπόν αυτό είναι το δικό μου το σκεπτικό. Ας ενισχύσουμε λίγο την διάσταση αυτής της υποψίας δηλαδή ότι θα πρέπει να υφίσταται μια υποψία προκειμένου να ε, προβαίνουμε στον έλεγχο και να μην γίνεται ένας γενικός έλεγχος. Ευχαριστώ κύριο Σαντόκτον τώρα. Ευχαριστώ τους ε, προέδρου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές ε, ε, για τη δουλειά που έχουν κάνει. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο το έργο δύο συνεισηγητών όταν έχουμε δύο συνεισηγητές που πρέπει να, δύο επιτροπές που πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους και αντιλαμβάνομαι βέβαια πως έχουμε 10.000 παραβάσεις με βάση τις διασαβήσεις οι οποίες ε, εντοπίζονται κάθε χρόνο και φτάνουμε σε ε, έως και 300.000 ευρώ ε, κατασχέσεις. Οπότε αυτό που χρειάζεται τώρα να κάνουμε είναι να προσαρμοστούμε στον ολοένα και καλύτερα προσαρμοσμένο τρόπο με τον οποίο δρούν οι εγκληματίες. Άρα λοιπόν εδώ πραγματικά αποτελεί το συγκεκριμένο ζήτημα προτεραιότητα και η έκθεσή μας προσπαθεί να, να δώσει την καλύτερη, να απευθυνθεί, να ασχοληθεί καλύτερα με αυτό το ζήτημα και σε αυτό συμβάλλει και η διεύνηση του όρου της έννοια των διαθεσίμων, αλλά θα πρέπει να είμαστε ε, προσεκτικοί και πρόσωπο εδώ του ΕΛΚΕ νομίζω πως είχε δίκιο. Δηλαδή θα πρέπει να ε, ε, έχουμε και τι δυνατότητε να επιτρέπουμε σε εκείνου που μεταφέρουν νομίμω αυτά τα αριστά διαθέσιμα να το πράττουν και στο μέλλον. Οπότε αυτό που ε, εμείς προσπαθούμε εδώ να κάνουμε είναι πάντοτε να εντοπίζουμε εκείνους οι οποίοι παρανόμως προσπαθούν να να εξάγουν ε, στα διαθέσιμα και αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει από αυτούς τους νέους ε, κανόνες να υποφέρουν εκείνοι οι οποίοι νομίμως μεταφέρουν τα, στα διαθέσιμά τους και έχουμε ακούσει ιστορίες από κάποιους οι οποίοι νομίμως πράγματι προβαίνουν σε μια τέτοια μεταφορά. Εάν λοιπόν δούμε ε, καλές προτάσεις εδώ σίγουρα θα υπάρχει υποστήριξη από την πλευρά της πολιτικής ομάδας αλλά θα πρέπει να υπάρξει και σεβασμός στις αναλογικότητες. Για παράδειγμα όταν εαυτό μα ότι ενδεχομένω θα πρέπει να περιληφθούν στον ορισμό και προπληρωμένε κάρτε. Είναι κάτι τέτοιο πραγματικά αναλογικό. Δηλαδή οι εγκληματίε συχνά, επειδή ακριβώ δεν θέλουν να, να συλληφθούν, δεν μεταφέρουν οι ίδιοι αυτέ τι προπληρωμένε κάρτε. Οπότε ε, αυτή η προσθήκη ενό ορισμού για ασυνόδευστα λεφτά διαθέσιμα είναι πολύ χρήσιμο. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά το σχετικό όριο που θα εφαρμόσουμε σε ό,τι αφορά τι αξίε, πράγματι θα είναι και αυτό ενδιαφέρον ε, και υπάρχουν και σε ό,τι αφορά την περίοδο και τη διαβίβαση των πληροφοριών. Σίγουρα θα πρέπει να το συζητήσουμε και περαιτέρω και να φτάσουμε σε μια συμφωνία και όπως είπα δεν θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω άφθες για όσους μεταφέρουν νόμιμα τα λεφτά διαθέσιμα. Αλλά το κυριότερο πρόβλημα που εγώ εντοπίζω είναι κυρίως ε, θεσμικού αν θέλετε χαρακτήρα. Πρώτος διακόπτη μέχρι τη 1 και 10 θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει οπότε. Ναι. Ε, δύο λεπτά είχαμε τοσα στους ομιλητές. Καλώς ο πρόεδρε μπορώ πολύ σύντομα να ολοκληρώσω. Ζητώ συγγνώμη, δεν ακούσει ότι έχουμε μόνο δύο λεπτά χρόνο Άρα λοιπόν, οι αρμόδιες ε, αρχές εδώ ε, για τους χρηματοοικονομικούς ελέγχους ε, καλούν να υπάρξει μια κοινή ομάδα οικονομικών πληροφοριών, αλλά αυτή σίγουρα θα πρέπει να σέβεται την αρχή της αναλογικότητας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κ. Αρτόρ τώρα για την Άλντε. Ναι, μόλις είδαμε τι σημαίνει το να κλέβει κανείς τον χρόνο των άλλων. Ο μελητής. Πολύ σύντομος θα είμαι. Γνωρίζω πως είναι ε, δύσκολο να ασχοληθεί ε, κανεί ε, και να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Γιατί, για παράδειγμα, σε ένα κινούμενο σχέδιο μπορεί κανεί εύκολα να εντοπίσει τον ληστή, τον απαταιώνα, τον εγκληματία που φοράει μια μαύρη μάσκα οτιδήποτε. άλλο στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να τον εντοπίσουμε. Οπότε βλέπουμε εδώ την προσπάθεια που κάνουν οι συγητέ και οι Επίτροπη αντιμετωπιστεί ειδικότερα το ζήτημα ε, της ε, έλλειψης πληροφοριών και σίγουρα χρειαζόμαστε ε, εντατικότερη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων ομάδων οικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών και των χωρών και όλες οι προσπάθειες που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση για αυτή την επίτευξη της συνεργασίας είναι ευπρόσδεκτες. Προηγούμενοι ομιλητές αναφέρθηκαν στο ζήτημα των ασυνόδευτων ρευστών και εμεί είμαστε τη ίδιας άποψη εξετάζουμε και εμείς ε, την έκθεση αυτή την περίοδο με τον Γιάσερ και σε ό,τι αφορά και τις ε, τροπολογίες που θα υποβάλουμε και τα 15 δευτερόλεπτα, 15 δευτερόλεπτα που περισσεύουν τα χαρίζω σε εσάς, στους υπόλοιπους. Η ε, Μπάρβαρα Κάπελ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που πήρα και μερικά δευτερόλεπτα παραπάνω. Θα είμαι σύντομη. Τα περισσότερα υπόθηκαν. Σίγουρα το σχέδιο έκθεσης ε, θα βελτιώσει και θα συμπληρώσει με τους ορισμούς τον κανονισμό, τον κανονισμό 1898-2005. Χρειαζόμαστε σαφείς ορισμούς για να υπάρξει εναρμόνιση και για τις κυρώσεις και για την υποχρέωση δήλωσης. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η αρχή της αναλογικότητας. Αν τώρα διευρύνουμε τόσο πολύ τον ορισμό του ρευστού και σε διάφορα πολύτιμα αντικείμενα και μέχρι χρυσάφι, άμα έχεις ένα ακριβό ρολόι στο χέρι σου, που δεν ξέρει κανείς ποια είναι ακριβώς η αξία του. Θα πρέπει δηλαδή κυρίως να βασιστούμε όχι στην περισσότερη γραφειοκρατία, αλλά να έχουμε καλύτερους ελέγχους βασιζόμενοι στον καθορισμό του ποιος είναι ύποπτος πριν αρχίσουμε τους ελέγχους. Πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα όπου υπάρχει υψηλή πιθανότητα να κάνουμε ελέγχους. Όπου δεν υπάρχει υψηλή πιθανότητα να είναι ένοχος ε, κάποιος, να αποφεύγονται οι ελέγχοι. Περισσότερη αρμόνιση χρειάζεται, καλύτερη έλεγχη των διαφόρων ειδών ε, χρηματοδότησης ρευστό της τρομοκρατίας. Όλα αυτά θα υποστηρίζουμε και ευχαριστώ πολύ. Η Άννα Γκόμες. Η πραγματική πρόκληση θα είναι η εφαρμογή. Και θα είναι σοβαρή η εφαρμογή. Τα κράτη-μέλη λένε το PNR είναι πολύ σημαντικό μέσο κατά καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Αλλά ξεχάσανε τα ιδιωτικά αεροσκάφη. Το περισσότερο χρήμα που ξεπλένεται από τους κλεπτοκράτες στην Ευρώπη μπαίνει στα αεροδρόμια μας μέσω ιδιωτικών αεροσκαφών που δεν τα ελέγχει κανείς. Οπότε, άκουσα ότι δεν έχει συμπεριληφθεί στην οδηγία η αποστολή ποσών μέσω ταχυδρομικών πακέτων. Όπως η Western Union για παράδειγμα. Μιλώντας με τις πορτογαλικές αρχές μαθαίνω ότι αυτοί τους ανισχούν, η Western Union. Συμπεριλαμβάνεται ή όχι. Και τέλος. Ελέγχει κανείς ότι οι ελεύθεροι λιμένες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής αυτών τον κανόνα που αποφασίζουμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Δύο λεπτά για τους ε, μας. Τελικές παρατηρήσεις. Και οι δύο θέλετε το λόγο, ωραία. Ωραία, τότε να αντιστρέψουμε τη σειρά. Ντελβό. Προς διευκρίνηση. Τα κοσμήματα δεν καλύπτονται από τη σχετική διάταξη όσα ρόλεξ θέλετε πάρτε μαζί. Γιατί στο παράδειγμα υπάρχει ο σχετικός ορισμός του ισοδυνάμου ρευστού Για την Άννα. Όχι δεν υπάρχει γι' αυτό που ρώτησε η υποχρέωση δήλωση. Και αυτό και συζητήθηκε. Οι περισσότεροι είχαν πει στη ζήτηση ότι δεν θέλουν να προβλέπετε αυτή η υποχρέωση δήλωση για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Για τα πακέτα. Από ό,τι γνωρίζω, τα τελωνία έχουν αρμοδιότητα να ελέγχουν τα ιδιωτικά αεροσκάφη. Ε, βέβαια και υπάρχει πρόβλημα με το bitcoin και τους εγκληματίες που το χρησιμοποιούν, αλλά δεν έχει υλική υπόσταση και άρα δεν μπορεί να κρυφτεί από τον κανονισμό. Δεν αποτελεί ρευστό. Ξανά ευχαριστώ για την καλή συνεργασία με τους κοιόδες Λόπες Αγγίγια. Πάρα πολύ σύντομα. Ακριβώς όπως είπε η συνάδελφος. Η Ντελβό λάβαμε υπόψη όλα τα λογικά αιτήματα των σκιοδοχέ βέβαια και μας προβληματίζει το τι επιπτώσεις θα υπάρχουν για τον Κοσμάκη που δεν θα πρέπει χωρίς καμία διάκριση να είναι αντικείμενο υποψιών. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ακριβής ρύθμιση. Είπαμε όχι στα προσωπικά αντικείμενα όπως κοσμήματα και ρολόγια και τις συνήθεις αποσκευές που πέραν από το τελωνίο, αλλά θα πρέπει το νομοθέτημα να εστιαστεί σε μεγάλα ποσά, τα οποία πρέπει να δηλωθούν στο χρυσό. Συζητήσαμε για τις προπληρωμένες κάρτες ενδελεχώς και μακροσκελώς και είπαμε ότι υπάρχει κατάχρηση αυτών. Διότι κατά κόρον χρησιμοποιούν για να παρακάμψουν τα όσα σήμερα ισχύουν. Έτσι κι αλλιώς έχουμε περιθώριο αλλαγών προσεχώς και είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε, να καλύψουμε όλα τα αιτήματα των συναδέλφων όσα είναι λογικά και να καταλήξουμε σε κάποιους συμβασμούς. Άρα ολοκληρώσαμε. 25 δεκάτος στις 3 ώρα είναι η προθεσμία. Δύο Νοεμβρίου θα τη συζητήσουμε και θα γίνει η ψήφιση της Επιτροπής 4 δωδεκάτου. Ευχαριστώ τους από τις δύο επιτροπές και εσένα Ρομπέρτο θα συνεχιστεί η συνεργασία μας. Και η συνεργασία των σχεδόν με τους σκιώδες. Συνεχίζει τη συνεργασία της η στι 2 ώρα. Ευχαριστώ.